της ημερήσιας διάταξης για αυτή την εβδομάδα η διάταξη η οποία εγκρίθη με βάση το άρθρο 49 στις 19 Νοεμβρίου. Σας έχει διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη. Όσον αφορά τη σημερινή μέρα η ομάδα της Ενωμένης ΕΕ Αριστεράς ε, έχει ζητήσει επίσης σε προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νέα στρατηγική ε, ευημερία των ζώων επ' ε, όσον αφορά την καλή συμβίωση των ζώων. Θα ψηφίσουμε την Πέμπτη. Και όσον αφορά την προφορική αιτιολόγηση αυτής της ερώτησης, η συνάδελφος Άνια Χάνιεθαμ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύμφωνα με τον δανεισμό άρθρο 152 ζητώ από το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την ε, συζήτηση για την προφορική ερώτηση 141-2015 με, μια, με ένα ψήφισμα σε ό,τι αφορά την καλύτερη βίωση των ζώων. Η σημερινή ε, στρατηγική θα τερματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου και δεν δείχνει οποιαδήποτε ένδειξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει για την κατάρτιση νέας στρατηγικής. Αυτό είναι παράδεκτο. Υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει ένα σαφή οδικό χάρτη προς την κατεύθυνση αυτή. Αγαπητοί συναδελφοί και από τον συνάδελφο εκ μέρους του συναδελφού Φαν Εκ, σας ζητώ να υποστηρίξετε το ψήφισμα αυτό για την ολοκλήρωση της συζήτησης και αν πιστεύετε ότι τα ζώα έχουν σημασία τώρα είναι η στιγμή να το δείξετε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Ποιο τάσεται υπέρ αυτής της ερώτησης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την κυρία Χάζενκαμπ για την πρωτοβουλία που έλαβε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν πολλά νομοσχέδια και πολλή νομοθεσία η οποία έχει περάσει από το Κοινοβούλιο αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι συνεκτικά όμως, δεν αποτελούν μια συνολική στρατηγική, δεν αποτελούν ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Αυτό τι σημαίνει ότι υποφέρουν τα ζώα, σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες σε διάφορες χώρες και ότι δεν έχουμε σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα, μια πραγματικά ενιαία αγορά. Άρα υποστηρίζω την πρόθεση της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτή την πρόταση. Από ό,τι βλέπω όχι. Μισό λεπτό. Εσείς διαφωνείτε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύγκριση. Ε, η μία ομάδα ζήτησε να υπάρξει ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τις τρομοκρατικές ενέργειες και ρωτήσαμε την Επιτροπή τι θα κάνει για να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα μέτρα που εγκρίθηκαν και που δεν είχαν ε, μπει στην πράξη και θα μπορούσαν να σώσουν εκατοντάδες ζωές. Με εκπλήσει λοιπόν το Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρίνουμε ότι ένα ψήφισμα για την ευζοία των ζώων ε, πάει ε, πάει μπροστά, είναι εμπροστοφυλακή έναντι ενός ψηφίσματος κατά της τρομοκρατίας. Κυρία Αλιού Μαρή, σας συγχαίρω γιατί με πολύ ε, καλή διατύπωση κατ' ουσίαν είσαστε υπέρ της αίτησης ε, ενώ πιστεύω ότι θελήσετε να μιλήσετε κατά αυτής. Ε, θα ψηφίσουμε όμως τώρα έτσι κι αλλιώς. Όποιος είναι υπέρ αυτής της πρώτης, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι συνάδελφοι επιθυμούν ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η πρόταση. Για την τρίτη δεν έχω προτάσεις ε, για την Τετάρτη η ε, ομάδα των Πρασίνων ζητάει την ψηφορία της έκθεσης Φερέρα Τόιρα σχετικά ε, με τα φορολογικά ειδοποιητήρια και καλ, μας καλεί να μεταφερθεί αυτή η ψηφορία για την Πέμπτη. Το λόγο έχει ο κύριος Λάμπερτς. Μιλήσαμε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της βελτιστοποίησης ε, των ε, εταιρικών ε, φόρων. Σήμερα εγκρίναμε την πρώτη έκθεση της, της Επιτροπής που δημιουργήθηκε ειδικά γι' αυτό. Έχουμε την εξή ανησυχία. Την προηγούμενη εβδομάδα η διάσκεψη των Προέδρων με πλειοψηφία αποφάσισε να αναβάλει για μία εβδομάδα την ε, ενδεχόμενη παράταση της Επιτροπής ΤΑΞ που αποτέλεσε αντικείμενο συνένεσης των πολιτικών ομάδων. Γιατί δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι θα εγκρίνουμε την έκθεση και μετά θα παρατείνουμε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμβαδίσουν οι δύο αποφάσεις. Στο μεταξύ, έλαβα σαφή μηνύματα από τις πολιτικές ομάδες, από την πλειοψηφία που είναι υπέρ της παράτασης. Η διάσκεψη των Προέδρων ενδεχομένως θα αποφασίσει την Πέμπτη και το θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια την Πέμπτη στις 12. Τότε εκλείπει το πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εγκρίνουμε την έκθεση την Τετάρτη και να ψηφίσουμε την παράταση την Πέμπτη υπήρχε μια αμφιβολία στην ε, προηγούμενη διάσκεψη των Πρόεδρων, αλλά ε, εάν έτσι κι αλλιώς παραταθεί η, ζωή της Επιτροπής τάξη, τότε δεν υπάρχει λόγος να παρατείνουμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάμπερτς. Ο κύριος Ντεμάζη θέλει να ταχθεί υπέρ της αίτησης, υπέρ της πρότασης αυτής. Κύριε Πρόεδρε, πριν από ένα περίπου χρόνο με τα LuxLeaks ε, εμφανίστηκαν αυτές οι σκανδαλώδεις συμφωνίες ε, με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυεθνικές με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να κλείσει ε, μια υπόθεση πριν υποβληθούν τεκμήρια και αποδείξεις. Εμάς όμως δεν μας δώσανε την πρόσβαση στα έγγραφα. Στο Κοινοβούλιο αυτό είναι γνωστό, υπήρξαν πολλές διαπραγματεύσεις Γι' αυτό λοιπόν εγώ κάνω έκκληση να αναβάλλετε τη ψηφοφορία, πέστε το ενδιάμεση έκθεση με οτιδήποτε άλλο. Η εντολή δεν μπορεί να εκπνεύσει. Πρέπει να αναβληθεί το θέμα αυτό, να αλλάξει η μερίσια διάταξη, γιατί αλλιώ θα είμαστε παντελώ αναξιόπιστοι όσον αφορά τον αγώνα μα κατά των φορολογικών παραδείσων. Ο κύριο Βίμπα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κάποια εξήγηση. Ε, εγώ από ό,τι είπε ο εκπρόσωπος των Πρασίνων κατάλαβα ότι ότι θα αποσυρθεί η πρόταση εάν τελικά στην Ολομέλεια ταχθούμε όλοι υπέρ της παράτασης. Και θέλω να σας πω ότι το ΕΛΚ επιθυμεί την παράταση των μηνών ακριβώς για να διαλευκανθούν τα θέματα τα οποία εκκρεμούν. Άρα ε, δηλαδή αν ε, το επιβεβαιώσουν αυτό και άλλες πολιτικές ομάδες θα ταχθούμε όλοι υπέρ της αναβολής της ψηφοφορίας την Τετάρτη. Κάπως έτσι το κατάλαβα και εμείς σας επαναλαμβάνω ως πολιτική ομάδα επιθυμούμε να διαλευκανθούν ε, τα θέματα που εκκρεμούν. Ο κύριος Ζήμων, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Όσον αφορά τους ε, σοσιαλδημοκράτες, ε, θέλω να σας ανακοινώσω ότι ακριβώς επειδή έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η αναταραχή, οι σοσιαλδημοκράτες υπέρ της ψηφορίας ε, την Τετάρτη Φεραίρα, την Πέμπτη στη διάσκεψη των Προέδρων και την Πέμπτη το μεσημέρι να ζητήσουμε την παράταση της ζωής της Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν είμαι ευγνώμων στον συνάδελφο κύριο Λαμπέρτ που αποσύρει την πρότασή του. Άρα δηλαδή αποσύρετε την πρότασή σας. Πολύ ωραία. Πρόεδρος. Κατόπιν τούτου δεν έχουμε άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη αυτής της εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατόπιν τούτου περνάμε στην κατάσταση πρόοδου της αναπτυξιακής ατζέντα της Ντόχα εν ώψη της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης. Και επ' αυτού έχει το λόγο καταρχήν η Επίτροπος η κυρία